Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αποτίσω τιμή σήμερα σε έναν μεγάλο άνδρα. Το Σάββατο Μισελ Ροκάρ ε, πέθανε στην ηλικία των 85 ε, ετών και ο παλαιός μας ε, ε, συνάδελφος είχε επιδείξει μεγάλο ζήλο και από το 1994 ως το 2009 είχε συμμετάσχει στις εργασίες και είχε επιδείξει ότι το Κοινοβούλιο και τα μέλη του δεσμεύονται με σταθερή προσήλωση για μια δίκαιη υπόθεση στην υπηρεσία των πολιτών. Ε, θυμάμαι πιο προσωπικά από τον ε, ακάματο Μισελ Ροκάρ, του οποίου το γραφείο ήταν δίπλα στο δικό μου, ε, πρώην ε, Πρωθυπουργό, ο οποίος ε, είχε, εργάστηκε σαν απλός βουλευτής και πραγματικά θα και τους συναδέλφους με τη δική του εργασία και την προσωπικότητά του πριν γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Επιτροπής Πολιτισμού. Η Γαλλία πραγματικά από όλες έναν μεγάλο Ευρωπαίο και έναν μεγάλο μίζωνα πολιτικό. Και θυμόμαστε για τις ε, συμφωνίες του Μαντινιό, οι οποίες επέτρεψαν να εξευρεθεί μία λύση όσον αφορά τις βιοπραγίες στη Νέα Καλλιδονία. Ο ζήλος του για την, υπερσπέρασπιση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του Αρκτικού Πόλου και της Ανταρκτικής, επιβεβαιώνει την υψηλή του ποιότητα ως οραματιστού. Ε, και θα του θα τιμή ε, την Πέμπτη ε, και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να γερθούν ούτως ώστε η δική μας συνέλευση να αποτίσουν τιμή στο Μισελ Ροκάρ σήμερα. je vous remercie. Πριν ε, κηρύξω την άνοιξη